όμως απαγορεύτηκε το δικαίωμα των βουλευτών να καταθέσουν τροπολογίες. Υπάρχει ένσταση σε αυτό που δεν απαντήθηκε. Η νομική υπηρεσία η ίδια ε, απεφάνθη θετικά υπέρ του δικαιώματος κατάθεσης των τροπολογιών. Η νομική υπηρεσία και η Επιτροπή ΑΦΚΟ έπρεπε να γνωμοδοτήσουν και αυτό δεν επετράπει. Ε, κατετέθησαν τροπολογίες οι οποίες απερίφθησαν. Αυτή η ε, ε, αντιμετώπιση στην έκθεση Εστρέλα αντίκειται στον κανονισμό και στην γνώμη της νομικής υπηρεσίας όπως παρουσιάστηκε στην Επιτροπή και εκφράζω τη σοβαρότατη ένστασή μου δεδομένου ότι είναι ευαίσθητο το θέμα που οδήγησε σε διαδηλώσεις ε, πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα με το οποίο προς, γίνεται προσπάθεια να καταπιεστεί μια πρωτοβουλία των πολιτών που συγκέντρωσε ένα εκατομμύριο υπογραφές. Ε, διαμαρτύρομαι έντονα απέναντι σε αυτήν την άκρος αντικανονική ε, στάση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. ναι, έλαβα και μια επιστολή σχετικά από δέκα συναδέλφους, η οποία όμως απαντήθηκε. Οπότε η κριτική της μη απάντησης δεν μπορεί να αναφέρεται σε μένα αλλά σε κάποιον άλλον. Επίσης η διάσκεψη των Προέδρων ενημερώθηκε ε, για τις ε, επί της ουσίας ενστάσεις σας. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να, ε, θέσει, να αφήσει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της αυριανής ημέρας. Ζητεί άλλος παρακαλώ τον λόγο για τη την ημερήσια διάταξη της σημερινή. Αποφασίσαμε λοιπόν σχετικά με την ημερήσια διάταξη και την διάταξη των εργασιών. Αρχίζουμε λοιπόν την κοινή συζήτηση για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Καταρχήν τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, κοινή αλλιευτική πολιτική. Η συγκίτρια κυρία Ρόντου